Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Άρχεται εκ νέου συνεδρίαση, κυρίε και κύριοι. Έχει μου μοιραστεί τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και σα παρακαλώ να μου δηλώσετε αν υπάρχουν αντιρρήσει. Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη έχει τώρα πέντε ψηφίσματα για το Ιράν, για τη Σιρήν Εμπαντή και δίνω το λόγο στον κύριο Ματσάκη. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε που μόλι φτάσατε, η δίωξη τη κυρία Σιρήν Εμπάντη, βραβείου Νόμπελ, είναι